Good afternoon, ladies and gentlemen. Please be so kind to take your seats. I know that today is 20th of July. It's vacation time, but... Γεια σας κυρίες και κύριοι, καθίστε. Ξέρω ότι σήμερα κανονικά πρέπει να είναι αργή, αλλά τι να κάνουμε, αυτή είναι η τιμή, το τίμημα της επιτυχίας, ότι πρέπει να είμαστε εδώ και να εργαστούμε. Είναι λοιπόν μεγάλη μου τιμή το ότι προεδρεύω αυτής της συνεδρίασης, ούτως ώστε να μπορέσουμε να δούμε τι θα κάνουμε για το άξιμο του Προέδρου της Επιτροπής Δημοσιονομικού Ελέγχου. Οπότε σας προτείνω την εξής ημερησία διάταξη. Πρώτον, έναρξη συνεδριάσεως. και ορισμός του προσωρινός προεδρεύοντος. Δεύτερον, διαδικασία. Την θα εκλεγεί ο πρόεδρος, επίσης θα εκλεγούν οι αντιπρόεδροι στη συνέχεια διάφορα και πέμπτον ανακοίνωση της επόμενη μας συναντήσεω. Συμφωνείτε με αυτή την ημερησία διάταξη. no Δεν βλέπω να υπάρχει καμία ένσταση, οπότε αφού δέχεστε συμφωνείτε με την ημερησία διάταξη, τότε συνεχίζουμε. Our list of Do we have quorum to make a decision. Θα πρέπει να αποφασίσουμε επομένω πώ για τη διαδικασία. Many members who have present, the quorum is eight. Νομίζω ότι η απαρτία είναι 8. Πόσο έχουμε.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 Η δήλωσή σα. θα ήθελα να σας πω ότι ο παλιό καταγό αναφέρει τον κύριο Φαντεκάμπ ότι αυτό θα μας εκπροσωπήσει εμά του Ολλανδού, όμω αλλάξαμε τι θέσει μα, και επομένω ε, λέει η κυρία Ντελάνγκε, εγώ θα εκπροσωπήσω του Ολλανδούς και όχι ο κύριο Φαντεκάμπ. Και θα έρθει σε 10-15 λεπτά. Όχι, όχι, τον αντικαθιστώ, παίρνω τη θέση του, το ρόλο του σε αυτή τη συνεδρία. So uh, our sitting is able uh, to make a decision. Let me... Ναι, αλλά πρέπει κάτι να αποφασίσουμε. Λοιπόν, θα είμαι σαφέστατος. Σκοπός είναι η εκλογή του Προεδρίου της Επιτροπής, δηλαδή του Προέδρου και των Αντιπροέδρων, ε, αν δεν απατώμε. Ο αριθμός των Αντιπροέδρων αποφασίζεται αποφασίζεται τώρα. Yes, Τέσσερις θα έχουμε. Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ζητήσω να γίνει μυστική ψηφοφορία. Ε, με συγχωρείτε, αλλά έχω μετάφραση, ρωτάει ο Πρόεδρος. Η κυρία Γκρέσλε ζητά ε, μυστική ψηφοφορία. Για όλο το Προεδρείο, παρακαλώ, θα ήθελα μυστική ψηφοφορία. Λοιπόν, ποιος είναι υπέρ της ε, αιτήσεως της ε, κυρίας ε, Γκρέσλε για να ψηφιστεί όλο το Προεδρείο με μυστική ψηφοφορία. Κυρία Γκρέσλε. Εάν ένας το ζητά, κύριε Πρόεδρε, απλώς υιοθετείται η πρόταση. Ευχαριστώ. Οπότε θα, εκλέξουμε τώρα το Προεδρείο. Θα ξεκινήσουμε με την ψηφοφορία για τον Πρόεδρο της Επιτροπής. Ευχαριστώ. Σύμφωνα με τον κανονισμό αν υπάρχουν πολλοί υποψήφοι, από ό,τι μου λέει η γραμματεία μπορούμε να έχουμε μυστική ψηφοφορία. Εάν τουλάχιστον ε, το ζητήσουν έξι μέλη της Επιτροπής. Πρέπει λοιπόν να δούμε αν υπάρχουν έξι μέλη της Επιτροπής που συμφωνούν να γίνει μυστική ψηφοφορία. Ποιος είναι υπέρ της μυστικής ψηφοφορίας. Δεκατέσσερις. Εφόσον είναι 14 υπέρ, υπέρ του να έχουμε μυστική ψηφοφορία, ποιος είναι κατά. Ε, Τρει κατά. Οπότε θα προχωρήσουμε με τη μυστική ψηφοφορία. Και αυτό θα ισχύσει για όλο το Προεδρείο. E, λοιπόν, ξεκινούμε με τον Πρόεδρο. Οπότε ε, πρώτα απ' όλα όμως χρειαζόμαστε ψηφολέκτες, αλλά ο κύριος Χατζημαρκάκης έχει ζητήσει το λόγο. Θα ήθελα να κάνω μία ε, ε, πρόταση. η κυρία Γκρέσλε προτείνει να γίνει μισική ψηφοφορία και για τον πρόεδρο. Εγώ προτείνω τον κύριο Λουίτζι Ντεματζίστης σαν υποψήφιο για την Προεδρία. Ευχαριστώ. Λοιπόν, αυτό είναι ε, υποψηφιότητα για την Προεδρία. Υπάρχει άλλος υποψήφιος για την Προεδρία της Επιτροπής. Δεν βλέπω άλλον, αλλά ο κύριος Οντή ζητά το λόγο. Κύριε Πρόεδρε, ρωτήσατε αν υπάρχει και άλλη ε, άλλη υποψηφιότητα. Ήθελα να ξέρω εάν υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι ήδη έχουν σεβαστεί τις προθεσμίες και έχουν υποβάλει υποψηφιότητα. Μπορούμε και σήμερα να αποφασίσουμε. Κύριε Δεμαγκίστρης, ο κύριος Δερμαγίστρης υπέβαλε την υποψηφιότητα του εχθές, το οποίο ήταν εντός των προθεσμιών για την ανακοίνωση των υποψηφίων. Κοιτάζοντας την αίθουσα, Υπάρχει καμία επιθυμία ο κύριος Χατζημαρκάκης υποστηρίζει έναν υποψήφιο ο οποίος όμως είναι ο μόνος υποψήφιος για την Προεδρία της Επιτροπής. Αντιλαμβάνομαι ότι δεν υπάρχουν άλλοι υποψήφοι. Εφόσον λοιπόν δεν υπάρχουν άλλοι υποψήφοι, μπορούμε να κλείσουμε τον ε, κατάλογο των ε, υποψηφίων για την ε, Προεδρία. Κυρία Γκρέσλε, κατόπιν αυτού, εφόσον δεν υπάρχει άλλος υποψήφιος πρόεδρος, επιμένετε να υπάρξει μυστική ψηφοφορία για αυτήν την θέση. Ωραία τότε χρειάζεται να εκλέξουμε ψηφολέκτες. και αυτό καλύπτεται από τον κανονισμό και λέγεται εάν, εάν ένας ένας μόνο υποψήφιος υπάρχει μπορεί να γίνει διαβοής. Να προχωρήσουμε διαβοής. Λοιπόν, έχουμε μυστική πληροφορία, έναν υποψήφιο, κύριε Ντεμαγκίστρης, δέχεστε να αναλάβετε την ε, θέση αυτή. Εντάξει. Οπότε, τώρα χρειαζόμαστε τα ονόματα των ψηφολεκτών, δύο ψηφολέκτες υποψηφίους. Κυρία Γκρέσλε, έχετε να μας προτείνετε ε, ε, ε, ψηφολέκτες ή να τα τραβήξουμε κλήρο. Εγώ θα πρόστινα την κυρία Κιώσσελα και τον κύριο Ιτέλε. Λοιπόν, τότε θα τραβήξουμε κλήρους. Ο κύριος Γκέμπεν Βάντεν Μπράντε. και ο κύριος Μάρτιν Έρενχάουζερ. Δύο ψηφολέκτες νομίζω αρκούνε. Θα πρέπει οι ομάδες να μας πούν επίσης ε, ε, ποιοι από τους ε, αναπληρωματικούς έχουν δικαίωμα ψήφους. Αυτό πρέπει να το πούν οι πολιτικές ομάδες. Με συγχωρείτε, αλλά δεν νομίζαμε ότι θα έχουμε μυστική ψηφοφορία. Λοιπόν, μέχρι να οργανώσουμε τον κατάλογο ψηφοφορίες θα, ε, θα πρέπει οι συντονιστές να μας πούν ποιοι θα εκπροσωπήσουν τις ε, πολιτικές ομάδες χωρίς ε, να μην ξεπερνούν ε, οι ψήφοι τις θέσεις για κάθε πολιτική ομάδα και χρειάζεται να ξέρω ποιοι θα είναι ε, μέλη της Επιτροπής και ποιοι αναπληρωματικοί. E για το ΕΛΚ. Ποιος ψηφίζει σαν αναπληρωματικός για το για το ΕΛΚ. Έχετε 11 υποψηφίους, δηλαδή μπορείτε να έχετε 11 ψήφους. Παρακαλώ αποφασίστε και πέστε μας ποιοι θα ψηφίσουν αν δεν παρήσανται όλοι. Δέκα από τα μέλη μας είναι παρόντα, ένα μέρος δεν είναι παρόν και παρακαλώ τον κύριο Βολμάιερ να ψηφίσει ως αναπληρωματικός. Και στη θέση, ποιον αντικαθιστά ο κύριος Βολμάγερ. Τον κύριο Ρεβελίνη. Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Πόσα, μέλη έχουμε στην ε, ομάδα. Λοιπόν, έχουμε 7 παρόντες μέλη. Το, οι φιλελεύθεροι. Ο κύριος Χατζημαρκάκης. Πράσινη 2. Ο κύριος Στάς. ECR, ε, κύρια Τσέσκοβα και ο κύριος Σαρνέσκι. Ε, Συντηρητική, δύο. Ε, έχετε δύο πλήρη μέλη ή υπάρχει και κανείς αντικαταστάσεις. Δεν έχετε αντικαταστάτες. Ε, γκουε, αριστερά. Ο κύριος Σόντεργαρτ, ένας. Ε, η EFD ένας ε, μόνος και από τους ανεξαρτήτους ο Μάρτιν Έλερ Χάουζερ παρίσταται. Δηλαδή έχουμε τώρα το κατάλογο των ποιοι, ε, αυτών οι οποίοι δικαιούνται να ψηφίσουν. Λοιπόν, σας υπενθυμίζω ότι εφόσον έχουμε έναν αντιπρόσωπο, ένα μόνο υποψήφιο, θα πρέπει να λάβει την πλειοψηφία των ψήφων που θα υπάρχουν ε, στην κάλπη. Με αυτόν τον τρόπο θα προχωρήσουμε, είναι μια διευκρίνηση. Τώρα άλλο τεχνικό θέμα, παρακαλώ τα μέλη της Επιτροπής και τα αναπληρωματικά να σηκώσουν το χέρι τους για να ξέρουμε σε ποιους θα πρέπει να δώσουμε ένα χαρτάκι για την ψηφοφορία. Ένα ψηφοδέλτιο. Και ένα ψηφοδέλτιο για μένα επιπλέον παρακαλώ κύριοι.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 Λοιπόν, θα διαβάσω τώρα όλα τα ονόματα και παρακαλώ όσοι ακούν το όνομά τους να έρχονται να ψηφίσουν. And Marta Andreasen, are you ready, ready to vote? Marta Andreasen, κυρία μου είσαστε έτοιμοι να ψηφίσετε, σας περιμένουμε.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 Andreasen, are you Κυρία Αντρεάσεν, ετοιμαστήκατε. Και ο κύριος Σαν Πιέρ Όντι να ετοιμάζεται. Ines Αιάλα Σέντερ.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 Andra Czeszkova. She is absent and no substitute. Hadzimar Kakis. Andra Cozzolino. Ryszard Czarnecki.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 Γκίλε Ιταλά. Καταλίν Ιβάν. Ιλιάνα Ιβάνοβα. Elisabeth Kostinger. Monika Luisa Makowej. Jan Olbrycht.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 Mr. Lefort instead of. Oui, oui. Theodoros Skylakakis. Soren Zondergaard. Bart Stas. Georgios Stavrakakis and Bogusław Liberacki. Scrutators, we need probably six and a half minutes to make these countings. Θα χρειαστούν ε, λίγα λεπτά οι ψηφολέκτες και θα έλεγα για 6-6,5 λεπτά να διακόψουμε τη συνεδρίαση αλλά μην βγείτε από την, ε, από την αίθουσα. Oh, excuse me. Your substitute, Paul.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

Μην πάτε μακριά σας παρακαλώ. Εδώ κοντά κοντά. Ladies and gentlemen. Κυρίες και κύριοι μου, παρακαλώ προσοχή. Θα ήθελα να ανακοινώσω τα αποτελέσματα. Εψήφισαν 28. Έλαβαν. Ναι, 25, όχι 3 απόλυτη πλειοψηφία 15 ο κύριος Λουίτζι Ντεμάγκιστρης είναι πρόεδρος της Επιτροπής μας. Congratulations. Welcome. Συγχαρητήρια, παρακαλώ ελάτε εδώ να λάβετε το έδρανο και να κάνετε τη δουλειά σας να... Πριν αρχίσουμε πρώτα πρώτα να ευχαριστήσω την πολιτική μου ομάδα η οποία με όρισε ως ε, υποψήφιο για την Προεδρία. Επίσης θα πρέπει όσους με υπερψήφισαν να τους ευχαριστήσω. Είναι πάρα πολύ σημαντική στιγμή για μένα. Πάρα πολύ σημαντική πολιτική εμπειρία. Θα έχω πάρα πολλά να μάθω από τους ε, παλαιότερους εδώ, αυτούς που ήδη διετέλεσαν ευρωβουλευτές. Θα επιστρατεύσω θέληση, ενθουσιασμό και θα επιστρατεύσω όλες τις επαγγελματικές γνώσεις για το έργο αυτής της Επιτροπής. Έχω διατελέσει σαν αρκετά χρόνια και νομίζω ότι αυτό θα βοηθήσει τη δουλειά μας ε, εδώ. υπάρχει αμοιβαίος σεβασμός και πιστεύω ότι θα μπορέσει ο καθένας εδώ να κάνει ό,τι πρέπει. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντική η λειτουργία του έργου επιτελεί αυτή η Επιτροπή. Είναι θέμα της διαφάνειας. Είναι θέμα του να εξασφαλίσουμε το ότι ε, όλα θα γίνονται όπως πρέπει, όλα γίνονται σύνομα, ιδίως όσον αφορά τις σχέσεις μας με τα άλλα θεσμικρόνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιστεύω ειλικρινά ότι βρισκόμαστε σε πάρα πολύ σημαντική συγκυρία και ε, μιλώντας για ε, διαφάνεια, αυτό σημαίνει ότι όλοι θα πρέπει να κάνουν αυτό που πρέπει, αυτό θυσμένο, θα πρέπει να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των Ευρωπαίων προς το Κοινοβούλιο. Και ε, αν ρίξουμε μια ματιά στα όσα παράτυπα ή παράνομα συμβαίνουν, ε, δική μας δουλειά είναι να τα προλαβαίνουμε. Είναι να στείλουμε ένα μήνυμα του ότι όποιος σέβεται τα συμπεφωνημένα θα έχει καλύτερη αντιμετώπιση του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιο και αντίθετα όποιος ε, παρεβαίνει και υπερβαίνει τα σκαμμένα αυτός θα τιμωρείται. Οπότε, σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά που με υπερψηφίσατε και ε, συγγνώμη αν τυχόν σας φαίνεται η περιβολική, η συναισθηματική μου φόρτιση. Τώρα, θα προχωρήσουμε στην εκλογή του πρώτου αντιπρόεδρου της Επιτροπής μας. Θα ήθελα τώρα να δω ποιοι είναι οι υποψήφοι. Do atto che è pervenuta una lettera del segretario generale del gruppo EFD che candida eh, l'onorevole Marta Andreasen come primo vicepresidente della Commissione. πρώτη αντιπρόεδρο. Δεν ξέρω αν υπάρχει τώρα κάποια άλλη πρόταση. Ε, κάποια πολιτική ομάδα ή κάποιο ατομικά θέλει να ζητήσει και για αυτή την ε, ψηφοφορία να γίνει διεξαγωγή. Μίστηκα. Ιδάλλω ε, θα ψηφίσουμε διαβοή. Ε, έχει κάποιος κάποια ένσταση. Θέλουμε μυστική ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Herr Präsident, ich möchte für unsere Gruppe erklären, dass wir den Antrag auf geheime Abstimmung unterstützen. Κύριε Πρόεδρε, υποστηρίζουμε το αίτημα αυτό για μυστική ψηφοφορία και από την ομάδα μας. E θα δούμε, θα δούμε. Νομίζω όμως ότι υπάρχει ο απαραίτητος νενομισμένος αριθμός η απαρτία που απαιτείται για μυστική ψηφοφορία. Για να τους μετρήσουμε όμως ψηλά τα χέρια σας, όλοι όσοι θέλετε μυστική ψηφοφορία. Μάλιστα, υπεραρκή. υπεραρκή. Για τον πρώτο αντιπρόεδρο λοιπόν θα χρησιμοποιήσουμε μυστική ψηφοφορία και θα είναι οι ίδιοι οι δύο ψηφολέκτες εκτός αν έχετε καμιά αντίρρηση οι ίδιοι. Παρακαλώ όσοι θα ψηφίσουν για τον πρώτο αντιπρόεδρο να σηκώσουν το χέρι και θα τους δώσουμε τα ψηφοδέλτια.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 αν υπάρχει κανένας αναπληρωματικός που θα ψηφίσει μαζί με τα πλήρη μέλη. Πρόεδρε, εσείς θα ψηφίσετε, παρακαλώ επιβεβαιώστε ότι θα ψηφίσετε. Εσείς, Πρόεδρε, θα ψηφίσετε. Io no, voto No, ha chiesto se lei ha l'intenzione di votare. Io no. No, al posto mio c'è il Α, εγώ όχι. Ο αναπληρωτής μου Χρήστος Ντέιβις. Bei uns fällt Prego, onorevole Gas. Ja, bei uns fällt wieder Frau Hohlmeier. Dankeschön für den Kollegen Rivellini. Dankeschön. Κυρία Χολμάγερ θα αντικαταστήσει και πάλι όπως πριν τον κύριο Ιβανίνη.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 L'onorevole Ines Ayala Sender. L'onorevole Zigmantas Balcitis. L'onorevole Andrea Cescova.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 Onorevole Tamas Deutsch. L'onorevole Martin Ernauser. Onorevole Jens Geier.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 Itala, si legge. Big Itala. Onorevole Vil Itala. Onorevole Sorin Catalin Ivan. Liliana Ivanova. Onorevole Elisabeth Kostinger. Onorevole Boguslav Liberadski. Onorevole Luisa Monica Macovei. Onorevole Jan Olbricht.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 Onorevole Teodoros Skilakakis. Onorevole Bo Soren Sondergaard.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 η ψηφοφορία των επομένων ε, υποψηφίων αντιπροέδρων διαβοή. Ε, έτσι καλώς πρέπει να φύγουμε, γιατί έχουμε υποχρεώσει άλλε επιτροπέ και πρέπει λοιπόν πολλοί από τους αδέλφους μα να φύγουν. Συμφωνώ. Δεν βλέπω κανείς να έχει ε, αντίρρηση για δεύτερο, τρίτο και τέταρτο αντιπρόεδρο. Να δούμε τις υποψηφιότητες. Ποιος θέλει το λόγο για την θέση του δευτέρου αντιπροέδρου. Πρέγω, νωρίβολε γράφη. Ich schlage für unsere Fraktion Jean-Pierre Audi vor. Danke. Jean-Pierre Audi, εκ μέρους της γύρω μας πολιτικής ομάδας, λέει κύριε Γκάις. Consente la nomina. Consente la... Συμφωνείτε? υποψήφια. Ναι, λέει ο κύριο Σοντή. Αν δεν έχει κανεί ένσταση, τότε θα θεωρηθεί ω υποψήφιο για τη δεύτερη θέση και ψηφίζουμε διαβοή. Prego, invito a prendere posto alla Presidenza. Καλό, κύριε Αντιπρόεδρε, ελάτε να λάβετε θέση στη, στο στεδρόνο τη Προεδρία. Τρίτο υποψήφιο αντιπρόεδρο. Ποιο θα είναι για την Επιτροπή μας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εμείς προτείνουμε σαν τρίτο αντιπρόεδρο τον συνάδελφο Λιμπεράτσκι. Μπορούμε να προχωρήσουμε διαβοής στην ε, εκλογή του κυρίου Λιμπεράτσκι. Και lo invito anche a lui a prendere posto alla presidenza. Prego, onorevole. παίρνει για την τετάρτη αντιπροεδρία το λόγο η ομάδα. θα πάρετε το λόγο για την τετάρτη αντιπροεδρία. Αξιότιμε κύριε. Με συγχωρείτε. Ε, ε, προτείνω τον συνάδελφο Ούνανσφορ. Έχετε κάτι να πείτε. Νόμιζα ότι θέλετε να εγκαταλείψετε την Τετάρτη Αντιπροεδρία. Διαφορετικά ε, προτείνω το, στον υποψήφιο να έρθει να αναλάβει την, το κάθισμα του Τετάρτου Αντιπροέδρου. Σε αυτό το σημείο λύεται η συνεδρίαση. Θα ε, συνεδριάσουν στις 9 ε, οι συντονιστές, στις 10.30 όλοι οι υπόλοιποι. Άρα καλό απόγευμα.